Doamnă președintă! Uh, Καλησπέρα, συναδελφοί. Άρχεται η συνεδρίαση. Να σας ενημερώσω ότι τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης είναι πλέον διαθέσιμα.